Οι αρμόδιες ουγγρικές αρχές κάνουν ε, πρόταση για την άρση της ασυλίας του κ. Ιστβαν Ιουελχή στα πλαίσια ποινική διαδικασίας. Η πρόταση αυτή ε, αποστέλλεται σύμφωνα με τον κανονισμό στην